Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελπίζω ότι θα έρθουν και τα υπόλοιπα μέλη όπου να είναι. Ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη. Έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω. Έχω υπάρξει δύο αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει διανέμηθει. Η πρώτη αλλαγή είναι κάτι το θετικό η Προεδρία πρότεινε στο Συμβούλιο να κάνει μια συμβιβαστική λύση για το θέμα των φυσικών καταστροφών. Ανεπίσημες διαπραγματεύσεις είχαν ήδη δείξει ότι η συμβιβαστική η οποία είχε προταθεί θα μπορούσε να γίνει δεκτή από τα κράτη-μέλη και θα μπορούσε επίσης να στηριχθεί και από την πλειοψηφία των μελών της μας Επιτροπής. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους πήραν μέρος στην ανταλλαγή email. Μας έδωσε την δυνατότητα να στείλουμε το μήνυμά μας εγκαίρως στο Συμβούλιο. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν το Συμβούλιο απέστειλε τη συμβοβαστική του πρόταση επίσημα με τη μορφή της επιστολής που ε, υπέγραψε ο πρέσβης της Προεδρίας. Σας απεστάλλει από τη Γραμματεία την ε, Τετάρτη, 24 Μαΐου. Όλοι είναι ενήμεροι γι' αυτό. Θα πρέπει να το βάλουμε σαν δεύτερο θέμα προς ψηφοφορία. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς το κλείσιμο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας προτείνω λοιπόν να προσθέσουμε μια δεύτερη ψηφοφορία Α, αύριο το πρωί. Ευχαριστώ. Ο κ. Βανίστελ Ροϊ. Να ευχαριστήσω και εγώ, λέει ο κ. Βανίστελ Ροϊ, τα μέλη τα οποία πήραν μέρος στην προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Ε, εσείς είστε αυτοί που συνδύασε τις ε, δύο προσπάθειες και ψηφοφορίες, όχι μόνο το θέμα του Συμβουλίου και τη συγχρηματοδότησης από τη μία, αλλά και με την αλληλεγγύη από την άλλη, έτσι ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο δυνατό ποσοστό του 95%. Δεν είναι μια πρόσκληση για να βρούμε άμεσα χρήματα, αλλά είναι μια καλή συμβιβαστική πρόταση και νομίζω ότι τελικά βλέπει κανείς ότι το να εμένει κανείς στη θέση του είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο Συμβούλιο. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν και σας ευχαριστώ. Ναι, ε, νομίζω ότι έχουμε μια καλή συμβιβαστική πρόταση. Νομίζω ότι συναντηθήκαμε στα μισά του δρόμου η μεν και η δε. Ξέρετε ότι εμείς θέλαμε το 100% και με 5% όριο αλλά η θέση του Συμβουλίου ήταν 90% συγχρηματοδότηση χωρίς όριο. Ε, και οι δύο πλευρές λοιπόν δέχτηκαν κάπως να υποχωρήσουν και τέλος έχουμε τώρα πια τη λύση 95% και 100%. Ε, προφανώς δεν είναι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους συνομοθέτες και είναι και κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε γρηγορότερα με το θέμα των φυσικών καταστροφών και θα επιτρέψει επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν τις περιφέρειες οι οποίες έχουν χτυπηθεί από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, σαν παραδείγμα. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα μέλη που υποστήριξαν την διαδικασία Ελπίζω να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και την ψηφοφορία αυτή αύριο. Η δεύτερη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη είναι νέα. Ο εμπειρογνώμων, ο οποίος θα μας παρουσίαζε τα αποτελέσματα της μελέτης που ζητήσαμε για την τελευταία προγραμματική περίοδο, ο κύριος Φέριν, από το Πανεπιστήμιο του Στραφκλάιντ, δυστυχώς δεν είναι σε θέση να είναι μαζί μας αύριο το πρωί. είναι θύμα του χάους που έφυξε τους επιβάτες της British Airways, ε, ακυρώθηκε το αεροπλάνο του και δεν μπορεί να βρει έγκαιρα άλλη πτήση. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε εδώ εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν συμφωνείτε μπορούμε να κρατήσουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη και να γίνει η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Εντάξει. Ο κύριος Βανίστελροι. Υπάρχει κάποιο έγγραφο γύρω από αυτό το θέμα. Έχουμε ε, μία περίληψη ε, στο φάκελο που σας έχει δοθεί. Ο κύριος Βανιούτεμποργκ. Κοιτάξτε έτσι και αλλιώ θα γίνει η παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων και γι' αυτό θα προτιμήσω παρακαλώ να το συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες, να το αναβάλουμε το θέμα και όχι να το σπάσουμε ε, σε μία συζήτηση μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τότε οι εμπειρογνώμονες των πανεπιστημίων ε, γιατί έκαναν τις μελέτες που έχουν αναλάβει. Γι' αυτό παρακαλώ θα ήθελα να υπάρξει μια συνολική άποψη και να αναβληθεί η συζήτηση. Ο κύριος Βόγγν, μια ερώτηση. Η πρόθεσή σας είναι να προσκαλέσετε τους εμπειρογνώμονες σε μια μελλοντική συνάντηση. Φυσικά, μπορούμε, ναι, μπορούμε, λέει η Πρόεδρος, μπορούμε να προγραμματίσουμε τη συνάντηση αυτή στο μέλλον. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Καλώς. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχει η λογική, εφόσον μπορούμε να καλέσουμε τις εμπειρογνώμονες σε μια άλλη ημερομηνία, τότε θα αναβάλουμε τη συζήτηση για την επόμενη συνάντηση, για να έχουμε μια πλήρη συζήτηση μαζί τους. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Με αυτές τις αλλαγές παρακαλώ να δεχθείτε την ημερησία διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάποια άλλη ανακοίνωση να κάνω. Μία από τις ε, ανακοινώσεις θα μπορούσε να είναι η αντιπροσωπεία στις Ασόρες, αλλά ο κύριος Σόμερτζή δεν είναι μαζί μας σήμερα, οπότε η παρουσίασή του θα γίνει αύριο. Και τώρα λοιπόν θα φτάσουμε στο επόμενο θέμα. Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2018 όλα τα τμήματα να καλωσορίσω τον κύριο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας, ο οποίος είναι ο Γενικός Εισηγητής του Κοινοβουλίου για το 2018. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μουρεσάν είναι υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής που είναι το 95% του συνόλου προϋπολογισμού της Ένωσης. Συνεργάστηκε λοιπόν ο κύριος Μουρεσάν και επιθυμεί τη συνεργασία με τις διάφορες τομεακές πολιτικές. Ε, ο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Επιτροπής είναι οι περιφερειακές πολιτικές και γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και με χαρά σας έχουμε ανάμεσά μας σήμερα κύριε Μουρεσάν. Θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν την παρουσίαση της πρότασης προϋπολογισμού της Ένωσης από την Επιτροπή που θα γίνει αύριο. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να ακούσουμε τον κύριο Μουρεσάν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ και εγώ. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μία φάση της δημοσιονομικής διαδικασίας όπου σαν κοινοβούλιο Έχουμε υιοθετήσει την έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον επόμενο χρόνο. Την Ολομέλεια του μηνός Μαρτίου. Και αυτή είναι η έκθεση η οποία περιελάμβανε τις πολιτικές μας προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο. Συνέταξα εγώ την έκθεση η οποία έγινε δεκτή από μεγάλη πλειοψηφία της Ολομέλειας και λέει στην Επιτροπή αυτά τα οποία περιμένουμε εμείς από αυτήν σαν βασικές προτεραιότητες το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ επισκέπτομαι όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συζητήσω με τους συναδέλφους, για να τους παρουσιάσω γενικά το ποιοι είναι οι βασικοί τομείς επικέντρωσής μας για τα επόμενα χρόνια δημοσιονομικά και να ακούσω επίσης και από εσά να μου πείτε το τι είναι σημαντικό να κάνουμε και πράγματι οι αρμοδιότητές σας είναι σαφείς και ευρείες και θα ήθελα με ενδιαφέρον να σας ακούσω σήμερα. Θέλω η παρουσία μου εδώ σήμερα να είναι η αρχή της συνεργασίας μας, γι' αυτό και ήρθα νωρί, πριν παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της η οποία θα γίνει αύριο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις, να ξεκινήσουμε ένα κάποιο διάλογο, γιατί θα είναι σημαντικό και για μένα σαν γενικής, γενικός εισηγητής πριν από τις διαπραγματεύσεις με Συμβούλιο και Επιτροπή, να είμαι ενήμερος για το ποιες πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στους δικούς σας τομείς ευθύνης. Δύο θέματα αυτή τη στιγμή εξελίσσονται. Πρώτον, συζητώ με όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και δεύτερον, Αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2018. Εμείς λοιπόν θέτουμε τις προτεραιότητές μας. Αύριο η Επιτροπή θα κάνει τις προτάσεις της. Θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών καταρχάς και μετά το Κοινοβούλιο θα καθορίσει την θέση του. Μετά θα την στείλουμε στο Συμβούλιο και στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, η λεγόμενη συνδιαλλαγή, και φυσικά όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα συντάξουν γνωμοδοτήσεις τις οποίες θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη. Τώρα σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο. Εγώ έχω δύο καταρχάς προτείνει, δύο τομείς στους οποίους πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Πρώτον, ανάπτυξη θέσης εργασίας και δεύτερον, ασφάλεια, λειτουργική και απλή ασφάλεια του πολίτη. Λοιπόν, ανάπτυξη από τη μία χονδρικά και ασφάλεια από την άλλη. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Πρώτον, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρώτον αυτό το οποίο απαιτείται έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, να, πρέπει να είμαστε ισχυροί οικονομικά. Πρέπει να είμαστε ελκυστικοί για τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως τις μικρομεσαίες, γιατί εκεί συνήθως δημιουργούνται οι θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν οι υποδομές όπως ε, το Connecting Europe, το Horizon 2020, οι μικρομεσαίες με το πρόγραμμα COSME, είναι σημαντικότατα προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω επίσης τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Η ανεργία των νέων είναι υψηλότατη στην Ευρώπη. Από την άλλη είμαστε ανοιχτοί στις παρατηρήσεις τις οποίες έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο τι λέει. Προσπαθώντας να θέσουμε σε λειτουργία την διευκόλυνση αυτή το μέσο αυτό πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να συνεχίσει τη λειτουργία του το μέσο αυτό, αλλά και να βελτιωθεί από τα μαθήματα που πήραμε τα τελευταία χρόνια. Το Erasmus επίσης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε γιατί δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για φοιτητέ, αλλά οι έρευνε δείχνουν ότι το 64% των εργοδοτών εκτιμούν την διεθνή εμπειρία που αποκτά κανείς όταν προσλαμβάνουν νέους. Η συμμετοχή λοιπόν στο Εράσμους δεν είναι μόνο ένα απλό πρόγραμμα ανταλλαγών, αλλά είναι κάτι το οποίο αυξήνει τις δυνατότητες τους να είναι επιτυχή στην αγορά εργασίας και είναι κάτι το οποίο διευκολύνει τελικά την κινητικότητα της εργασίας γιατί όταν έχει κάνει κανείς τέτοιου είδους προγράμματα Εράσμους γίνεται πιο ανταγωνιστικός να βρει δουλειά ακόμα και σε άλλη χώρα. Τώρα για την ασφάλεια και τη λειτουργική ασφάλεια. Οι πόροι τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας, τα τμήματα 3 και 4 είναι ιδιαίτερως περιορισμένοι. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους ελάχιστους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι υπηρεσίες της Ένωσης που έχουν ευθύνες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και νομίζω ότι με αρκετά λίγα χρήματα μπορούμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας και ταυτόχρονα να προωθήσουμε την ασφάλεια, τη λειτουργική ασφάλεια, την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Θέλω το ΕΑΣΟ, η Interpol, η Europol, η Eurojust ε, να μπορέσουν να αυξήσουν και τους προϋπολογισμούς τους αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και θα ήθελα επίσης να δω οι υπηρεσίες αυτές να συνεργάζονται καλύτερα. Υποστηρίζω επίσης και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για την άμυνα, τις οποίες πρόθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Υπάρχουν κάποιες οικονομίες κλίμακας στον τομέα της έρευνας στην άμυνα. Και αν πράγματι θέλουμε να κάνουμε κάτι στην άμυνα σε επίπεδο ευρωπαϊκό λόγω των οικονομιών κλίμακας, αντί να δαπανούμε τα χρήματα αυτά 28 φορές σε 28 χώρες, μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα άπαξ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μοιράσουμε τα ωφέλη σε όλες τις χώρες. Και φυσικά και μέσω ΝΑΤΟ και το να κάνει φυσικά κάτι για την άμυνά της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίφαση με το τι κάνει σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ε, το ΝΑΤΟ μάλιστα υποδέχεται θετικά τις ενέργειες αυτές σε σχέση με την ασφάλεια και τη λειτουργική ασφάλεια του πολίτη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στα πλαίσια της νότιας και ανατολικής γειτονίας. Θα είμαστε ασφαλείς στις κατοικίες μας αν έχουμε γύρω μας χώρες οι οποίες είναι όσο πιο ευημερούσες και ασφαλής γίνεται. Και γι' αυτό πολλές χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεση όπως η Γεωργία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες αυτές που είναι σημαντικές για το ευρωπαϊκό μέλλον και οι οποίες έχουν μπροστά τους μια όλο ένα πιο δραστήρια ρωσική ομοσπονδία. Και το ίδιο συμβαίνει και με την νότια διάσταση. Η Ορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με το προσφυγικό επίσης και γι' αυτό τα χρήματα τα οποία δίδονται για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του προβλήματος της μετανάστευσης πρέπει να δαπανηθούν σωστά και είναι πιο πολιτικά θα έλεγα εύκολο να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς και πιο ασφαλές για την Ευρώπη. Αυτά τώρα για τις βασικές προτεραιότητες. Στις κατευθυντήριες γραμμές τώρα λέμε ότι η περιφερειακή πολιτική είναι το βασικό επενδυτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων είναι απαράδεκτες, είναι κάτι το οποίο φυσικά με ενοχλεί. Και πρώτον, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς εσάς από πλευράς μου, εάν πράγματι υπάρχουν νέοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δαπανίσουμε χρήματα κοινοτικά σε χώρους και τομείς στους οποίους δεν είχαμε προβλέψει το 2013 όταν προβλέψαμε και αποφασίσαμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις τρέχουσες διαδικασίες και αυτό είναι κάτι το απαραίτητο και για την πολιτική συνοχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης όπως επίσης και της παράνομης μετανάστευσης αλλά κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των υποεξέλιξη προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν και τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια της πολιτικής διαφορετικών πολιτικών, καινοτομία δικτύων, σημαντικών γενικά για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τώρα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης πέρυσι δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε οι πιστώσεις υποχρεώσεων στο πρώτο τμήμα, οι διαχειριστικές αρχές δεν είχαν διοριστεί ακόμα και οι ανάγκες δεν ήταν πάρα πολύ σημαντικές επιτόπου. Θα αλλάξει όμως η κατάσταση για τον προϋπολογισμό του 2018 γιατί αν τα προγράμματα δεν θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ταχύτητα τον πέμπτο χρόνο του δημοσιονομικού πλαισίου, τότε πότε θα είναι. Συνεπώς λοιπόν σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών έχουμε 459 ε, σε λειτουργία από 560 περίπου που έχουν πιστοποιηθεί. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε πάρα πολλές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Σουηδία, και υπάρχουν και χώρες όμως που δεν πηγαίνουν πολύ καλά, όπως η δική μου χώρα, όπου έχουμε ε, πραγματικά ε, προχωρήσει με πολύ αργή ταχύτητα. Μόνο δύο διαχειριστικές αρχές από τις δέκα έχουν πιστοποιηθεί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ε, πριν από το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε επιτέλους τα προγράμματα να αποκτήσουν ταχύτητα κρουαζιέρας από το 2018 και να υπάρχουν αρκετά χρήματα στον προϋπολογισμό στις πιστώσεις υποχρεώσεων, ε, πληρωμών, συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο μήνυμα από ε, το οποίο μπορεί να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μην είναι, υπε... να μην είναι εντάξει στις ταμιακές της υποχρεώσεις. Είναι πολύ καλό και για τους εμπλεκόμενους και για τους ωφελούμενους ε, και δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω πάλι σε επίπεδο απλήρωτων λογαριασμών. Είδαμε τι έγινε το 2014 2,3 δις χρωστάγαμε τότε, είχαμε αφήσει απλήρωτα, το 2014 όμως ήταν έτσι, το 2015 έφτασαμε τα 25 δις. Τώρα καταφέραμε να μειώσουμε λίγο τα καθυστερημένα, εν μέρη τουλάχιστον. Αλλά για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο ε, γιογιό το οποίο νιώσαμε τα τελευταία χρόνια, που να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το χρέος, Καλό είναι να προσπαθούμε εμείς να αυξήσουμε το ποσοστό απορρόφησης, γιατί το ποσοστό αυτό είναι απογοητευτικό σήμερα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν επιστώσεις πληρωμών για τα επόμενα χρόνια, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι στο τέλος της δημοσιονομικής αυτής περίοδου θα αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προβλήματα με αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Δεν θα είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε και μπορούμε να το αποφύγουμε μέσω χρηστής διαχείρισης και σωστού ε, προγραμματισμού. Αυτά έχω αγαπητοί πρόεδρε ε, και αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι το βασικό επενδυτικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, πολιτική μας υπεριφερειακή. Αυτή τη στιγμή έχει έτσι και αλλιώς υψηλή θέση στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει οι διαχειριστικές αρχές να πιστοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να υπάρξει ροή πιστώσεων. Σχετικά με τα πιλωτικά τώρα. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι εδώ ήταν πολύ δραστήριοι. Σε αυτό κατέθεσαν 13 προτάσεις πριν από την προθεσμία, την 3η Μαΐου, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα έστελνε στην Επιτροπή προϋπολογισμών, τα συγκεντρώσαμε, τα στείλαμε στην Επιτροπή για αξιολόγηση και η διαδικασία από εδώ και πέρα είναι πρώτον, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει την πρώτη εκτίμηση, την πρώτη αξιολόγηση, να βαθμολογήσει τα προγράμματα και δεύτερον θα δημιουργήσουμε ένα πακέτο προγραμμάτων το οποίο θα προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν επί τη βάση της αξιολόγησης της πρώτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ένα πιλωτικό πρόγραμμα πάρει α ή β, είναι πολύ πιθανό να χρηματοδοτηθεί του χρόνου. Αν έχει μικρότερο βαθμό, τότε θα είναι μάλλον πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθεί. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτιάξουμε ένα συνολικό πακέτο και να προωθήσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν πάρει πράγματι υψηλή βαθμολογία. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Ιδιαίτερα για το πώς έχει η κατάσταση, εσείς γνωρίζετε το τι συμβαίνει με τις πληρωμές και με τις διαχειριστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να παραμείνουμε σε στενή επαφή κατά τη διάρκεια της συνολικής δημοσιονομικής διαδικασίας, έτσι ώστε να είμαστε ενήμεροι για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο πλήρη και λεπτομερή παρουσίαση. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Θα αφήσω τον εαυτό μου για το τέλος. Είμαι συγγήτρια και ελπίζω και εγώ όντω ότι θα είμαστε σε στενή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ποιος πρώτος, κύριος Φανίστερα, όχι, ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να μιλήσω για τον προϋπολογισμό αυτό για το 2018. Και θέλω λοιπόν να διατυπώσω κάποιες παρατηρήσεις. Σύμφωνο ότι πρέπει να επιμείνουμε στον προπολογισμό αυτό για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία απασχόλησης, την βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτό αποτελεί την προτερότητά μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές με τις οποίες ε, βρίσκεται απέναντι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι να δούμε ποιο τμήμα των δαπανών ανταποκρίνεται σε αυτήν την πραγματική σημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία αύξηση των δαπανών, να δούμε πόση θα είναι αυτή η αύξηση για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Έπειτα για τον ορίζοντα 2020, το ίδιο και ο έρασμος είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Πρέπει να δώσουμε νέα όθηση στο πρόγραμμα αυτό, το έρασμος, και αυτό είναι σημαντικό και για τους εργοδότες, γιατί το έχουμε διαπιστώσει ότι οι εργοδότες πιστεύουν πως η συμμετοχή κάποιων στέρασμος είναι ένα συν. Επίσης, πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και να προσθέσουμε 25 εκατομμύρια για την εγγύηση που θα προσφέρεται. Εδώ λοιπόν θέλω επίσης να επιμείνω στο ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και ένα μεγαλύτερο αποθεματικό στον προπολογισμό. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράμε πολύ γρήγορα αν υπάρξουν νέες ανάγκες. Άρα αυτή η ευελιξία στον προπολογισμό μας πρέπει να ενισχυθεί. Ένα άλλο ζήτημα που απορρέει από την πρόταση αυτή τη δημοσιονομική για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι θα γίνει με το διοικητικό κόστος. Γιατί και το Συμβούλιο θα ήθελε να μειωθεί το διοικητικό αυτό κόστος, το κόστος διαχείρισης. Οπότε, εγώ θέλω να ξέρω συγκεκριμένα τι προβλέπετε. Για το 2018 δηλαδή, πόσο μπορούμε να μειώσουμε τις διοικητικές δαπάνες, το κόστος διαχείρισης. Από την άλλη χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στις υποχρεώσεις. Είναι κάτι σημαντικό. Αλλά πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να απαλλαγούμε και τις δύο επόμενες χρονιές. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Βόγαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Πυρίνσκι είναι ο σκιώδης εισηγητές από τους σοσιαλιστές, αλλά θα αργήσει, γι' αυτό μου ζήτησε αν μπορώ εγώ να μιλήσω εκ μέρους του. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις κατευθυντήριες γραμμές που μας παρουσίασε. Τον ευχαριστώ που ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας οι σοσιαλιστές, όπως και οι περισσότεροι πιστεύω ευρωβουλευτές εδώ, εκφράσουν ικανοποίηση για τόσο αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου η πολιτική συνοχής να πρικοδοτηθεί κατάλληλα για το 2018 και μετά. Και όπως και συγκεκριτής για τον προπολογισμό και εμείς πιστεύουμε ότι η περιφερειακή μας πολιτική είναι βασικό στοιχείο αν θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία στην Ευρώπη. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι είναι και πιο σημαντική πολιτική και η πιο ορατή αυτή που μπορεί να προβληθεί περισσότερο παντού σε όλες τις περιφέρειες. Και έτσι ο κόσμος καταλαβαίνει τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπει ότι τα προγράμματα στις διάφορες περιφέρειες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο. Οι επενδύσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβάλλονται περισσότερο. Τώρα, έχουμε πει ότι μέχρι τώρα η χρήση των κονδυλίων δεν είναι επαρκής. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην αρχή, στην εκκίνηση των προγραμμάτων. Δεν ξέρω. Πάντα γίνεται αυτό. Πάντα υπάρχει καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα για τον προπολογισμό. Πάντως βλέπουμε ότι ζητάει περισσότερες πληρωμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνοχή. Οπότε, όπως λέει και ο εισηγητής, αν δεν έχει επαρκείς πόρους ή πολιτική συνοχής, δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και πρέπει να είμαστε σκληροί. Άκουσα ότι από το 2013 και μετά Κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλο καυγά ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τι πληρωμέ. Κάθε χρόνο από τα 13 και μετά. Και αναρωτιέμαι αν φέτο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όπω ξέρουμε, δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η, συγγνώμη, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα τιμήσει τι υποχρεώσει του πια από εδώ και πέρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον έχει πάρει τι αποφάσει που έχει πάρει. Οπότε είναι μία μάχη που θα χρειαστεί να δώσουμε του επόμενου μήνε. Πάντως και ο εισηγητής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών πρέπει να δώσουν τη μάχη για τη συνοχή. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Περιφέρειες, ακόμη και η Ουαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο δικιά μου, δηλαδή εκλογική περιφέρεια, για τα επόμενα δύο χρόνια θα χρησιμοποιεί κονδυλία συνοχής. Οπότε είναι ζωτική σημασία να γίνουν οι πληρωμές κανονικά και στο μέλλον. Δεν θα είναι κάτι εύκολο, αλλά ήθελα να το επισημάνω αυτό και στην δικιά μα εισηγήτρια τη δικιά μας επιτροπής, δηλαδή για τον προπολογισμό, να φροντίσει αυτό να τονιστεί επαρκώ και να δώσουμε τον αγώνα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλου, αν μη τι άλλο, να δώσει αγώνα προκειμένου να πρικοδοτηθεί επαρκώ η πολιτική συνοχή. Ευχαριστούμε κύριο Στόμασιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. θα μιλήσω και εγώ για τον Σκιώδη. Γνωρίζομαι ότι είναι πολύ σημαντική απόφαση και εφαρμογή για τον προϋπολογισμό. Από το τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο κάναμε μια πρόοδο στα πλαίσια της περίοδου 14-20. Δεν θέλουμε να ε, επαναληφθούν τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν διαρθρωτικά πριν ε, εγκριθεί το καινούριο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημαντικά θέματα για την Επιτροπή μας, ε, αφού ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε μία ε, πολύ στεναρή άποψη. Καταρχήν ευχαριστώ που ήρθατε πριν παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός στην Επιτροπή Budget του προϋπολογισμού. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή Ρέτζι να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία πληρωμών και ε, υλοποίησης του προϋπολογισμού για το 2017. Έχουμε πολύ σαφή άποψη ε, για τον προϋπολογισμό αυτό και θα συνεχίσουμε το ίδιο και το 2019. Όπως ε, αναφέρθηκε ήδη από τους συναδέλφους, επιμένουμε οι κατευθυντήριες γραμμές που υποστηρίχθηκαν από το Κοινοβούλιο φέτος το Μάρτιο να ακολουθούνται στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 19 γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική συνοχή να ακολουθήσει όλες τις παρατηρήσεις που εμπεριέχονται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερον, να πω ότι ο προϋπολογισμός ε, στηρίζει τις προτεραιότητες ε, που αναδείχθηκαν και υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά συμφωνώ μαζί σας που λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε δύο γενικές κατευθύνσεις, ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια για τους πολίτες. Για το πρώτο μέρος ε, έχουμε πολιτική που στηρίζει ε, τους στόχους μας στα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τη διαδικασία και να αποτρέπουμε ε, τυχόν ε, ε, εκρεμείς πληρωμές όπως είχαμε το, τα προηγούμενα έτη. Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, ενδεχομένως επικίνδυνη συσσόρευση εκρεμών πληρωμών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ανταπόκριση για τις πληρωμές που ζητούνται τα κράτη-μέλη για να αποδειχθεί ο ρόλος της πολιτικής μας και η ικανότητα της Ένωσης ε, να ανταποκρίνεται σε όλες τις, τις υποχρεώσεις του προϋπολογισμού και αυτές που απορρέουν από συμφωνίες με τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τον προϋπολογισμό και να τον υλοποιεί με βάση τα αποτελέσματα. Υπογραμμίζω την σημασία της απλούστευσης των κανόνων. Έχουμε πολύ έντονη θέση εδώ στην Επιτροπή Ρέτζη για την απλούστευση και υπογρα... το υπογραμμίζομαι αυτό και στη γνωμοδότηση για το φάκελο του πολυνομοσχεδίου Omnibus που αφορά τις δημοσιονομικού τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και ρυθμίσεις 2014-2020. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Η κέρυες προτεραιότητες είναι η επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση με έξυπνε επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα, ε, καινοτομία και ανάπτυξη, μεγαλύτερη υποστήριξη βέβαια των ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζω τον ρόλο κλειδί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας, είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιηθεί η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης για την βελτίωση του προϋπολογισμού και της υλοποίησής του. Τέλος, επιθυμώ να υπογραμμίσω επίσης ότι η καλύτερη συνεκτικότητα, ε, η συμπληρωματικότητα χρειάζονται συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων ταμείων ε, που επενδύουν σε εθνικά προγράμματα για να προωθηθούν οι επενδύσεις. Πιο στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να αναλυφθούν για την καλύτερη ορατότητα των ΕΔΕΤ ε, σε έργα και ε, επενδύσεις από διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα ταμεία. Αυτή είναι η βασική γραμμή που θα ακολουθήσω στη γνωμοδότηση και ε, πιστεύω ότι μαζί με τους σκιώδεις θα καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Ο κύριος Βαν Νίστελρόι. Ναι, μετά τα συμπεράσματα των ε, συναδέλφων και τα δικά σας κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Καταρχήν μιλάμε για ευελιξία στον προϋπολογισμό και στις κατευθυντήριες γραμμές επίσης. Αν υπάρχει ε, ένα που αν υπάρχει ε, οποιαδήποτε δυνατότητα ε, αύξησης ευελιξίας, την κάναμε. Και βεβαίως θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν χωρίς να υπονομεύσουμε τις συμφωνίες στα κράτη-μέλη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκρίναμε τους κανονισμούς για τη μετανάστευση. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι καινούριο, πρέπει να προσθεθεί μια νέα γραμμή στον προϋπολογισμό. Και εσείς το είπατε πριν. Όλα εξαρτώνται από τους στόχους μας απασχόληση και ανάπτυξη, ασφάλεια για τους πολίτες. Όλα αυτά πρέπει να τα ε, συμπεριλάβουμε. Και η ανάδειξη αυτών των προτεραιοτήτων σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, χαίρομαι για τις παρατηρήσεις σας, διότι αν θέλετε να ενισχύσετε την πολιτική συνοχή θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει. Ε, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα κονδύλια από αυτό το ταμείο είναι σημαντικά για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας ε, και θα μπορέσουμε έτσι να ε, οργανώσουμε τις ικανότητες που υπάρχουν σε επίπεδο περιφερειών, πόλεων, για να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες πληροφορίας, επικοινωνίας, να εφαρμοστούν οι βιώσιμοι στόχοι κλπ. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και όπως είπατε επίση πολύ σωστά, θέλουμε να ενισχύσουμε το Horizon 2020. Ε, γνώση και καινοτομία. Ε, χρειάζεται όμως και ένας διάδρομος προσγείωσης ε, ο οποίος θα μας εξασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν οι καινοτομίες ε, ε, θα αυξηθούν οι εξαγωγές, θα έχουμε μεγαλύτερη απασχόληση και ανάπτυξη. Ε, αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε ως βασική υποδομή, σαν να είναι η τροχή ενός αυτοκινήτου ανεξάρτητα από τον κινητήρα του. Θα πρέπει λοιπόν να όλα τα, όλες οι συνιστώσεις να συνεργάζονται. Και χαίρομαι με αυτή την προσέγγιση σας χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Ε, ξέρω ότι είστε ειδικό. Κάτι που δεν καταλαβαίνω είναι το εξή. Άκουσα ότι στις διαπραγματεύσεις για το 2017 η, σφορά, η συνεισφορά των χωρών στον προϋπολογισμό μειώθηκε λόγω της βραδίας έναρξης. Αν δεν αλλάξουν υποχρεώσεις όμως, στο τέλος ε, θα υπάρξει συσσόρευση υποχρεώσεων, διότι δεν θα έχουν γίνει οι πληρωμές ή θα πρέπει να αναβληθούν για αργότερα και λόγω του Brexit έχουμε πολλά προβλήματα. Μπορεί λοιπόν να πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια σημεία. Πώς μπορούμε να προλάβουμε το πρόβλημα, δηλαδή ότι οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν στα πλαίσια του προϋπολογισμού να ε, εκτελεστούν. Αυτά είναι κάποιες ανησυχήσεις. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, εμείς ε, για την απόδοση αλλάξαμε το σύστημά μας. Έχουμε τώρα πληρωμές βάσει της απόδοσης, προσανατολισμένης με τις προϋποθέσεις εκ των προτέρων κλπ. Η 6% του προϋπολογισμού μας έχει δεσμευθεί στους φακέλους των κρατών μελών για να δαπανηθεί υπέρ αυτών που έφτασαν σε καλά αποτελέσματα. Αλλά υπάρχει κάτι παράδοξο εδώ. Είπατε, κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει πολύ καλά και στη διαχείριση και στις δομές αναφέρατε κάποιες χώρες, ενώ άλλες δεν έχουν προχωρήσει. Το 2018, 17-18, πότε θα κρίνουμε τα αποτελέσματα και γιατί περιμένουμε μέχρι το 2019 για να δοθούν τα χρήματα. Αυτό είναι γραφειοκρατία. Και δεν την καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτές οι χώρες που ανταποκρίθηκαν καλά και άρχισαν γρήγορα να υλοποιούν τα έργα, θα πρέπει να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να τα δαπανίσουν το 2018. Γιατί να περιμένουμε μετά τις εκλογές. Πρέπει να δώσουν πριν από τις εκλογές. Πρέπει να έχουμε την ισχύ να πάμε στον κόσμο και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Να πείσουμε αυτοί που τα πήγαν καλά, αυτοί που δούλεψαν σωστά θα πάρουν τα χρήματα. Το 6% είναι 21 δις που έχει μπει στην άκρη ε, στο φάκελο των κρατών μελών. Εμείς θα ε, προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ως προς αυτό τον κανονισμό. Ε, ήδη το έχουμε ενσωματώσει στα δομικά στοιχεία για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. κύριος κύριε Μάτο, όχι. Άλλος κανείς, όχι. Καλώς. Λοιπόν, κύριε Μουρισόν για να απαντήσετε παρακαλώ να σχολιάσετε. Ναι, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία στις διάφορες κατηγορίες και το διοικητικό κόστος. Προς το παρόν είμαστε στις πολιτικές προτεραιότητες, εξού και δεν υπάρχουν νούμερα ακόμα για τον προπολογισμό του 2018. Αύριο θα γίνει αυτό, όταν η Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού. Έχουμε υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές, έχουμε πει με λόγια που θέλουμε περισσότερα, που περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει περισσότερα χρήματα, αύριο θα ξέρουμε περισσότερα και από τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε για νούμερα. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια το 2018 θα εξακολουθεί να είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασίλειου, θα εξακολουθεί να έχει πλήρη δικαιώματα και αρμοδιότητες και ευθύνε και υποχρεώσεις, οπότε θα εξακολουθεί να υποφελείται από τα κονδύλια. Τώρα η μελλοντική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να μην επηρεάσει καθόλου τον προπολογισμό του 2018. Βέβαια βλέπουμε ήδη ότι έμεσα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε συμφωνήσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εμεί την κάναμε τη δουλειά μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό που δεν ήταν τέλειο για μα, ήταν όμω ένα καλό συμβασμό που εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο επίση έπρεπε να τον εγκρίνει, αλλά η σημερινή κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπλόκαρε στο Συμβούλιο τα πράγματα μέχρι τι εκλογέ του Ηνωμένου Βασίλειο, τον Ιούνιο δηλαδή. Εντάξει, μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 9 Ιουνίου, δεν είναι πρόβλημα. Δύο μήνες καθυστέρηση δεν θα μας δημιουργήσει επί τόπου μεγάλα προβλήματα, αλλά αν δεν γίνει η δημοσιονομική αυτή μεταρρύθμιση, τότε ναι. Γιατί οι προτεραιότητες για τον προπολογισμό του 2018 θα είναι διαφορετικές από αυτές που υποθέταμε το 2013. Δεν είχαμε προβλέψει τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση, το μέγεθος με τον οποίο μας έφτασε, δηλαδή το θέμα της τρομοκρατίας, της ασφάλειας λοιπά Δεν τα είχαμε δει με τον τρόπο που τα βλέπουμε σήμερα. Έπειτα η αναθεώρηση των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών θέλει να ενισχύσει τον ορίζοντα 2020 την διευκόλυνση για την Ευρώπη. Γι' αυτό εξάλλου δημιουργήθηκε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να αντικαταστήσει την πολιτική συνοχή. Πρόκειται για διαφορετική προσέγγιση από τις επιχορηγήσεις. Θέλει να στηρίξει και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται στην καινοτομία. Πολύ καλό, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά την πολιτική συνοχής. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι η μεταρρύθμιση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών είναι ζωτική σημασίας και είναι προ όφελο και του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί θέλουμε να βάλουμε περισσότερα χρήματα στον ορίζοντα 2020 και αυτός που υποφελείται περισσότερο από τον ορίζοντα 2020 είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχουν πολλά πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, αριστείας, οπότε για πολύ καλούς και σωστούς λόγους είναι οι κύριοι που υποφελούνται από αυτά, οι κύριοι δικαιούχοι. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση αυτή. Αν την μπλοκάρει το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε βέβαια οδηγεί σε αβεβαιότητα τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή για την επόμενη χρονιά. Έπειτα, ο κ. Φανίστερον αναφέρθηκε στην ευελιξία. Έχει δίκιο. Από την αρχή της περίοδου, κάθε φορά που υπήρχε κρίση, εμείς αντιδρούσαμε, αποφασίσαμε να δημιουργηθεί η ευκολία, η διευκόλυνση μάλλον με την Τουρκία για τους πρόσφυγες και μερικές φορές έρχεται το, έρχονται δημοσιογράφοι και λένε κάποια πράγματα και ενώ εμεί τα ξέρουμε διαφορετικά. Λοιπόν, είναι σωστό που το κοινοβούλιο παρεμβαίνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σταθερότητα και ότι η θέση μας που είμαστε υπεύθυνοι για τον προπολογισμό και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τα προγράμματα τα οποία ήδη ισχύουν να μην τεθούν σε κίνδυνο. Αναφέρθηκαν εδώ κατευθυντήριε γραμμέ πολλέ φορέ. Ε, λοιπόν, όλε τι συζητήσει που είχαμε μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ κατάλαβα ότι παίρνουν στα σοβαρά τι κατευθυντήριε γραμμέ που εμεί υιοθετήσαμε, ότι καταλαβαίνουν τι προτεραιότητές μα, α ελπίσουμε ότι αυτό θα το δούμε και αύριο στην παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού. Βέβαια, όντω οι κανόνε μερικέ φορέ είναι περίπλοκοι και μου το λένε οι δικαιούχοι συχνά και οι επιχειρηματίε το λένε σαν βάρο. Λένε ότι το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι κανόνε είναι τόσο περίπλοκοι. Και για το άλλο που είπε για τις πληρωμές και για τις υποχρεώσεις ο κ. Φανίστερο, για να αποφύγουμε τη συσσόρευση ε, υποχρεώσεων και οφειλών στο τέλος, είναι καλύτερη λύση είναι να έχουμε απορρόφηση, καλή απορρόφηση. Γιατί όσο πιο πολλές είναι οφειλές στο τέλος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι και ο πολιτικός κίνδυνος μετά το Μάρτιο του 2019, τα δύο χρόνια δηλαδή μετά το άρθρο 50, ε, τότε θα πρέπει να τακτοποιήσουμε πάλι τα πράγματα και να τηρηθούν πλήρως υποχρεώσεις των χωρών μελών μέχρι το 2020. Πάντως η απορρόφηση αρχίζει και αυξάνεται σε ορισμένες χώρες. Οι διαχειριστικές αρχές βέβαια δεν ε, έχουν οριστεί ακόμα σε μερικές χώρες. Σε άλλες χώρες υπάρχουν και λειτουργούν καλά. Συνολικά το επίπεδο είναι απογοητευτικό όμως. Και ο στόχος πρέπει να είναι διαχειριστικές αρχές να έχουν καθοριστεί παντού μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Σας ευχαριστώ πάντως για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας που έχω καταγράψει εδώ και θα τις πάρω μαζί μου και προσβλέπω και εγώ στη συνέχιση του διαλόγου αφότου παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε και να εργαζόμεθα για την ε, κοινή μας θέση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή Ρέντζη και καλή συνέχεια στην έκθεση, την έκθεσή σας. Και τώρα προχωρούμε και πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι μια γνωμοδότηση για τη συγκρότηση κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Ο κύριος Μπόγκοβιτς είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης και θα του δώσω το λόγο. Υπάρχει προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης που είναι η 1η Ιουνίου 2017. Δεν βλέπω να αντιδρά κανείς. Καλώς. Οπότε θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής της 20 Ιουνίου. Κύριε Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον ε, Μάιο του 2014, ο κανονισμός 560 του 2014 ε, συνέστησε της, ε, ε, τη την κοινή επιχείρηση που είναι μια ε, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ Ένωσης και Κοινοπραξίας Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων και σε μια δεκαετή περίοδο προβλέπονται 975 εκατομμύρια και 2,73 δις από τις επιχειρήσεις βιοπροϊόντων, βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Στο consortium ε, ε, δίνονται τα χρήματα και μετά μέρος αυτών των κονδυλίων ε, προωθούνται στις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Ε, τα επιλέξιμα κονδύλια επιλέγονται και δίδονται στις επιμέρους βιομηχανίες. Αυτό το σύστημα δεν ήταν αποτελεσματικό γιατί δεν ε, αξιοποιούνταν τα κονδύλια στην κοινή επιχείρηση και δεν μπορούσαν να επιστροφούν τα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν η σύμπραξη αυτή πρότεινε το καταστατικό να τροποποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο. Θα έπρεπε οι εταιρείε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να, χρηματοδοτούν απευθεία έργα και να τα χορηγούν στη σύμπραξη για τη λειτουργία τους. Ε, υπάρχει συμφωνία και από την ε, Κομισιόν, γιατί έτσι η χνηλασιμότητα θα είναι καλύτερη και οι εταιρείε θα μπορούν καλύτερα να παίρνουν τις αποφάσεις τους και οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στη, στη χρηματοδότηση. Εγώ συμφωνώ με την θετική αυτή τροποποίηση όπως είπα, οι εταιρείε θα δραστηριοποιηθούν περισσότερο μετά από την αλλαγή αυτή και οι εταιρείε θα πρέπει να παρέχουν όλη την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της σύμπραξης, αλλά και για τα ίδια τα έργα. Προτείνω λοιπόν η Επιτροπή Ήτρε, που είναι η καθήλυνα αρμόδια, να ε, πάρει τη γνωμοδότησή μας που θα είναι, όπου θα εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας. Παράλληλα προτείνω μαζί με την Επιτροπή Ήτρε να ε, προετοιμάσουμε μια δημόσια ακρόαση το φθινόπωρο φέτος και να καλέσουμε εκπροσώπους των βιομηχανιών βιοπροϊόντων, εκπροσώπους της Κομισιόν και άλλους εμπλεκομένους και έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα τα έργα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του τομέα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν οι πόροι από ορυκτά καύσιμα ε, από βιοπροϊόντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την κυκλική οικονομία που πρέπει να προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, και η κυρία Νταντσού από τους Σκιώδης. Ευχαριστώ. Προπούς εν κάδρου Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και στα προγράμματα Horizon 2020 που αποτελούν τμήμα των προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία 14-20 Στόχος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη αυτών των βιοβιομηχανιών. Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της λεγόμενης βιοοικονομίας και μπορεί να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην οικονομική ανάκαμψη κάποιων κράτων μελών και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο ευφυούς ανάπτυξης υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και να περάσουμε σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα μέχρι το 50. Όπως είπε ο κύριος Μπόγκοβιτς, έχουμε να κάνουμε με μια εταιρική σχέση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 3,7 δις, ανάμεσα στην Ένωση από τη μία και ένα κονσόρτιο με επιχειρήσεων από την άλλη, στοιχηματίζοντας στον μετασχηματισμό των ανανεώσιμων πηγών σε καύσιμο και σε οικολογικά προϊόντα. Νομίζω λοιπόν ότι η χρησιμοποίηση των λεγόμενων βιοδιηληστηρίων θα μπορέσουν να μειώσουν α, την εξάρτηση της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα και να βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τις αλλαγές της κλιματολογικές. Το 2017 27 αεροπορικές επιχειρήσεις δέχτηκαν να διασφαλίσουν 5.000 ε, πτήσεις χρησιμοποιώντας ε, ε, μείγμα ανάμεσα στην κυροσύνη και το εναλλακτικό καύσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να κατασκευαστεί το καύσιμο αυτό σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη και να απαιτείται στις προδιαγραφές του ΙΚΑΟ. Είναι μια λύση έτσι ώστε ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών καυσερίων. Μέχρι τώρα οι βιοβιομηχανίες είναι το 3% του ετήσιου κύκλου της βιοοικονομίας, αυτό το μισό δις. Ενώ μπορεί η βιομηχανία αυτή να δημιουργήσει μέχρι και 22 εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Θέλουμε να αναπτυχθεί λοιπόν και θέλουμε να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον παραδοσιακό τομέα της βιοοικονομίας. Η Ευρώπη έχει την κατάλληλη τεχνολογική βάση για να χρησιμοποιήσει το δυναμικό αυτό με σωστό τρόπο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύει διάφορες πολιτικές επιλογές για την εφαρμογή του προγράμματος στα πλαίσια του Horizon 2020. Στόχος μας είναι να έχουμε μια εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και για τις μεγάλες βιομηχανίες και γι' αυτό χρειάζεται μια στρατηγική για μια νέα πολιτική στην Ευρώπη. Συμφωνώ με το ότι το κόστος λειτουργίας της κοινή αυτής προσπάθειας θα πρέπει να καλυφθεί από άμεσες καταβολές της βιομηχανίας και όχι μόνο του ίδιου του συνόλου του κονσόρτιου. Είναι αλήθεια επίσης ότι υπάρχει μια σειρά βιομηχανικών τομέων που μπορούν να συνεισφέρουν και σε επιμέρους μεμονωμένα προγράμματα. Η λύση αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί στα πλαίσια της κοινή προσπάθειας της σχετικής με τα ακενοτόμα φάρμακα. Και γι' αυτό ε, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω μια τέτοια πρόταση. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη παρακαλώ κύριε Δεμάτο. Il partenariato pubblico-privato fra e Νομίζω ότι θα πρέπει η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να βοηθήσει το μείωση του κόστους της έρευνας και να διασφαλίσει επίσης επαρκείς χρηματοδοτήσεις για τους εργαζομένους. Η CSC μας λέει ότι μπορεί να συνεισφέρει η οικονομία στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Δεν θα πρέπει αυτό όμως να δημιουργήσει περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Νομίζω ότι κάποια τεχνικά θέματα θα πρέπει να λυθούν άμεσα και να βρούμε λύσεις οι οποίες να μην βλάπτουν το περιβάλλον. Βασικός στόχος της βιοβιομηχανίας είναι να υποστηρίξει την ανεξαρτησία της Ένωσης από ορυκτά καύσιμα. Εδώ έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει ε, οι αναλλακτικέ λύσεις να φύγουν το περιβάλλον. Οι προτάσεις του Συμβουλίου, τις οποίες ο εισηγητής μας λέει να στηρίξουμε, είναι βασικό πρότυπο στα πλαίσια του Innovative Medicine, κάτι το οποίο μας δημιουργεί αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της έρευνας. Εκτός λοιπόν από την δυνατότητα πληρωμής του Consortium προς τις επιμέρους επιχειρήσεις, να προβλεφθεί επίσης ε, ε, και άμεση καταβολή ποσών από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει την, την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Θα κάνω τροπολογίες στην πρόταση του Συμβουλίου γιατί οι προτάσεις αυτές δεν βοηθούν την ελευθερία της καινοτομίας και της έρευνας, την ανεξαρτησία μάλλον. Ο κύριος Βανίστελο έχει το λόγο. Ναι, θέλω και εγώ το λόγο, παρακαλώ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και θα αρχίσω με τις δικές σας ερωτήσεις. Είναι δύσκολο να την καταλάβει κανείς αυτήν την απορία, γιατί εδώ δεν πρόκειται για την ανεξαρτησία της έρευνας και της ανάπτυξης, πρόκειται για την χρήση της γνώσης στην Ευρώπη. Μπορείτε να έχετε χιλιάδες καθηγητές που να έχουν δεν ξέρω πόσα βραβεία και πένους κτλ. Αν η βιομηχανία όμως δεν χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση, τότε μένουμε πίσω. Μεγάλες επιχειρήσεις ε, πηγαίνουν και κάνουν την έρευνά τους σε άλλα σημεία του κόσμου, φτιάχνουν ε, συνθετικά πρώτα λοιπά Αλλού. Άρα το ερώτημα δεν είναι πώς το χρησιμοποιεί η βιομηχανία, αλλά το θέμα της συνεργασίας αυτής και πιστεύω ότι είναι ένα θετικό πλαίσιο να έχουμε την προσέγγιση αυτή που έχουμε. Το πιο σημαντικό όμως που βλέπω εγώ εδώ είναι η θέση των περιφερειών, η οποία ενισχύεται έτσι. Γιατί στην αρχή αυτά τα κονσόρτια δημιουργούνται μέσω του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρώτα βρίσκεις τα χρήματα και μετά, αν τα καταφέρεις, βάζεις και κάποια στο πρόγραμμά σου. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μεγάλη ευθύνη που έχουν οι εταίροι σε μια περιφέρεια, να ο κύριος Μπόκοβιτς τα ξέρει και από την Σλοβενία, αυτό σημαίνει ότι θέλεις την επένδυση που κάνεις σε ένα πρόγραμμα να σου αποδώσει κάτι. Λες, ε, συγχρηματοδοτώ και έτσι μπορώ να υποφεληθώ για το δικό μου τον κλάδο, για τη γεωργία, τα νέα υλικά, την ξυλία, οτιδήποτε. Συνεπώς, εγώ το βλέπω σαν αποκέντρωση της διαχείρισης. Και εδώ ερχόμαστε με τα περιφερειακά κονδύλια. Πρόκειται για περισσότερη δίκευση. Αυτοί που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτήν την βιομηχανία βιοπροϊόντων μπορούν να το κάνουν. Και συγχρόνως συνδέονται και με άλλους με τους οποίους μπορούν να μοιραστούν τη γνώση και έτσι να χρησιμοποιήσουν ακόμα καλύτερα και πιο γρήγορα αυτήν την οικονομία. Η περιφερειακή πολιτική, η περιφερειακή μάλλον επιτροπή λοιπόν πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να δώσει την άποψή της, να πει ότι πρόκειται για αποκεντρωμένη διαχείριση, ώστε να είναι περισσότερος ο κόσμος που καταλαβαίνει το τι γίνεται και αυτό μόνο θετικά μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Πέρυσι ήμουν στην Πρατισλάβα σε μια συνάντηση κυρίως για τις νέες χώρες μέλη και εκεί πολλές περιφέρειες είπαν ότι θέλουν να προσαρμοστούν σε αυτήν την βιομηχανία βιοπροϊόντων, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές αγροτικέ περιοχές. Και ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Δεν χρειάζεται κανεί να είναι σε μια μεγάλη πόλη για να συμμετάσχει. Άρα λοιπόν βοηθάμε τα πράγματα να προχωρήσουν και να γίνουν πραγματικότητα. Βάζουμε ρόδες στο κάρο, όπως είπε ο κ. Φανίστερο. Συνεπώς, ναι, χρειάστηκε συνεργασία με την Ήτρε. Σωστά το λέτε. Θα το συζητήσουμε και στους συντονιστέ φαντάζομαι, σε λίγο, για την επιθυμία των Πρασίνων να κάνουν έκθεση διές πρωτοβουλίας. Πάντως αυτό το οποίο αφορά τόσες περιφέρειες πρέπει να βρεθεί και στην καρδιά οποιασδήποτε τέτοιας έκθεσης. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Αν λοιπόν έχουμε μια ακρόαση ή μια έκθεση βία πρωτοβουλίας, θα πρέπει να σταθεί πολύ κοντά σε αυτήν την οικονομία που βασίζεται στις βιομηχανίες βιοπροϊόντων. Δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια, πρόκειται και για νέα υλικά που βασίζονται στα βιοπροϊόντα. Κατευθείαν από φυτά, χωρίς να χρειαζόμαστε πια τα ορυκτά. Πρόκειται επίσης για βιοδιαχείριση. Υπάρχουν τρεις πυλώνες, σε αυτήν την ε, βιομηχανία βιοπροϊόντων. Ο Τραμπ το τελευταίο Σαββατοκύριακο τι είπε, είπε ας κάνουμε χωρίς το Παρίσι, χωρίς συμφωνία, τη συμφωνία αυτή των Παρισιών. Και τα σχόλια της κυρίας Μέρκελ χτες ήταν ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται ότι συνδυάζουμε τη γνώση, την επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή όλων στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σημαντικό τρίπτυχο για τα επόμενα χρόνια. Οπότε ίσως δεν ξέρω αν απαντάει και στην απορία σας. Μην το αμβλύνουμε έτσι, μην πέφτουν οι φιλοδοξίες μας, αντίθετα να ενισχυθούν. Πρόεδρος, υπάρχουν άλλοι από την Επιτροπή μας που θέλουν το λόγο, παρακαλώ, άλλοι ευρωβουλευτές, όχι. Ωραία, θα δώσω τότε στο λόγο, το λόγο στον κύριο Βάλντε Μαρκότ που είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητέ τον κύριο Ποκόβονετς και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και του κύριου Φανίστερόι που είναι ένας από τους πατέρες, θα έλεγα, της πρωτοβουλίας αυτής που ήταν εισηγητής πριν από μερικά χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν που αντιλαμβάνεστε την επιχειρηματική πραγματικότητα της πρωτοβουλίας αυτής. Οι αλλαγές που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ μικρές επιτρέπει στην βιομηχανία όχι μόνο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική πτυχή, αλλά και κατευθείαν σε προγράμματα. Κάτι είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για τεχνικής φύσεως τροπολογίες και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Θέλω επίσης να στηρίξω και κάποια από τα σχόλιά σας όσον αφορά για την αξία της ε, οικονομίας αυτή των βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Ενισχύονται όντω οι περιφέρειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίζουμε. Η οικονομία αυτή που βασίζεται στα βιοπροϊόντα είναι περιφερειακής φύσεως. Βιομάζα, είτε πρόκειται για τα απόβλητα, είτε πρόκειται για άλλες πηγές, χωματερές, Τα ωφέλη από τη βιομηχανία αυτή είναι τοπικά, οπότε ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι και θα το έχετε δει και στη Γερμανία. Η στρατηγική η σχετική με την βιοοικονομία έχει ανανεωθεί και στην Ιταλία και αλλού. Πολλές χώρες μέλη αντιλαμβάνονται ότι αυτή η βιοοικονομία έχει τη δικιά της αξία. Είτε πρόκειται για την κυκλική οικονομία, και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια. Πράγματι, οι βιομηχανίες που βασίζονται στα βιοπροϊόντα χρησιμοποιούν οποιοδήποτε πόρο για, για να χρησιμοποιηθούν στα λιπάσματα, για παράδειγμα. Παίρνουμε πρωτεΐνες από τέτοιους πόρους και επίσης χρησιμοποιούμε υλικά για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια πλαστικά από αυτά τα δύο προϊόντα. Πάντα λοιπόν μπορεί να υπάρχει βιοδηληστήριο που μπορεί να βοηθήσει να παρθούν 5-6 διαφορετικού είδους προϊόντα. Άρα λοιπόν συνεισφέρει η βιομηχανία αυτή δύο προϊόντων και στην ε, κυκλική οικονομία. Αυτές οι μικρές αλλαγές θα τη βοηθήσουν να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα από ό,τι λειτουργεί τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε E, Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων είναι πολύ σημαντικές και στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς. Είναι πολύ σημαντικές γιατί μπορούν να αλλάξουν τις ε, πηγές ε, ορεικτών καυσίμων σε άλλες πηγές. Δεν μπορούμε βέβαια, ε, επίσης δεν μπορούμε να μεταφέρουμε μεγάλες ποσότητες σε μεγάλες αποστάσεις. Και αυτός είναι ένας λόγος για αυτή την αλλαγή. Τη διαδικασία μπορούμε να την απλουστεύσουμε. Κάποιοι εμπλεκόμενοι έχουν συγκεκριμένα έργα και δεν θέλουν να παρεμποδιστούν από διοικητική γραφειοκρατία. Και εμείς έχουμε τον ίδιο στόχο και χαιρόμεθα που συμπίπτουν οι απόψεις μας. Ήδη έχουμε θέσει την προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Η Επιτροπή Ήτρε είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς θα ετοιμάσουμε την γνωμοδότηση, αλλά όπως είπα θα ήθελα να οργανώσουμε ένα hearing, μια ακρόαση για να συζητήσουμε τις κοινέ προκλήσεις που τόσο σημαντικές είναι για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα αξιοποιήσουμε την ε, δυνατότητα για την ακρόαση. Είναι πολύ σημαντικό και ε, θα... Ε, είναι σημαντικό και για τις περιφέρειες θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν αφορά μία, δύο, δέκα ή είκοσι βιομηχανίες. Είναι μια ευκαιρία οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι πόροι, να είναι προβληματικοί, αλλά μπορεί να γίνουν πόροι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιφερειακή ανάπτυξη και συμφωνώ με τις απόψεις που εκφράστηκαν εδώ. Ευχαριστώ και σας για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ήδη 1η Ιουνίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και στις 20 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και θα υποβάλλουμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ τη γνωμοδότησή μας. Το επόμενο θέμα είναι ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Επίτροπο ΣΥΜ Κάλλας για να δούμε αν έχει φτάσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σιμ Κάλλα, πρόεδρο της ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση για τους δικαιούχου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ΕΔΕΤ. Η ομάδα συστήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και πρόκειται για την ομάδα 18 εμπειρογνωμόνων ανεξάρτητων που θα εκτιμήσουν τα ΕΔΕΤ. Το καθήκον της ομάδας είναι να συμβουλεύσουν την Επιτροπή σχετικά με την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού βάρους. Η ομάδα συναντήθηκε 9 φορές πρόσφατα στις 16 Μαΐου και θα συναντηθεί άλλη μία φορά στις 11 Ιουλίου. Στις συνεδριάσεις μέχρι τώρα η ομάδα εξέτασε πολλά θέματα της απλούστευσης, για παράδειγμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απλουστευμένα κόστη, πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και τα χρηματοδοτικά μέσα, ο κανονιστικός υπερθεματισμός, ο έλεγχος, ε, βελτίωση της επιμερισμένης διαχείρισης, ενιαίοι κανόνες για τα ταμεία. Στην τελευταία συνάντηση θα εξετάσει τις συστάσεις για την πολιτική μετά το 2020. Η ομάδα είχε πρόεδρο έναν πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σιμ Κάλλας, ο οποίος ήρθε νωρίς ε, στην Επιτροπή μας το Φεβρουάριο του 2016 όταν άρχισε να συνεδριάζει τις πρώτες φορές η ομάδα αυτή και χαίρομαι που ξαναήρθε για να μας ενημερώσει για το έργο της, του της ομάδας καθώς τελειώνει το έργο αυτό. Και θα μας πει ε, κάποια πράγματα σχετικά με το τι θα αναμένουμε ως προς τα συμπεράσματα της, της ομάδας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σιμκάλας και μετά στα μέλη για ερωτήσεις και σχόλια. Και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καρποφόρα συζήτηση. Κύριε Κάλλας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία, τη δυνατότητα που μου δίνεται να συζητήσω αυτό το σημαντικό θέμα. Πριν από δύο χρόνια συμφώνησα να προεδρεύσω στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση, που είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα όπως ξέρετε. Και αυτό το έκανα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, πιστεύω στην επιμερισμένη διαχείριση και την πολιτική συνοχή έχουν προστιθέμενη αξία διότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και πράγματι έδωσαν ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα τις τελευταίες ε, δεκαετίες και μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω επίσης ότι το, το γραφειοκρατικό, ο γραφειοκρατικός φόρτος ε, δεν είναι αναπόφευκτος, ενώ τώρα τον συνδέουν οι πολίτες και οι δικαιούχοι με τα προγράμματα. Η ομάδα μας αποτελείται από 12 ανεξάρτητους υψηλού επίπεδου ειδικού με μακρά εμπειρία σε επιτυχείς διαχειριστικές αρχές, εταίρους, ε, αστικές ε, ε, δομές που γνωρίζουν πώς λειτουργούν στην πράξη οι αρχές μας. Και βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι σαν εμένα, πρώην μέλη της Επιτροπής και μέλη επίσης της ε, ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θυμάμε θυμάμαι ότι εντατικά συζητούσαμε για αυτά τα θέματα και τότε. Αυτή, αυτό το ποικίλο υπόβαθρο νομίζω ότι βοηθεί τους εμπειρογνώμονες να υποβάλουν ρεαλιστικές και συγκεκριμένες συστάσεις πάνω στη βάση καλής γνώσης του τι πήγε και τι δεν πήγε καλά κατά το παρελθόν. Ε, θέλουμε επίσης να αλλάξουμε το πολιτικό αφήγημα και να βοηθήσουμε να ε, υπάρξει ξανά εμπιστοσύνη ε, μεταξύ όλων των μερών σε εθνικό, ε, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο που παίζουν ρόλο για τα κονδύλια και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και την επιτυχία του εν συνόλο. Όλο και όσο πιο πολύ συζητούμε λεπτομερή θέματα, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η ρίζα του κακού. Μέχρι τώρα πολύ συχνά, αντί να πιάνουμε τη ρίζα του κακού, ε, των προβλημάτων, ε, προσπαθήσαμε να ε, λύσεις. Θέλαμε να κινηθούμε με κατευθυντήριες γραμμές, σε κάθε περίπτωση. Τώρα στη συνοχή έχουμε πάνω από 600 σελίδες νομοθεσίας στην επίσημη εφημερίδα και πάνω από 5.000 σελίδες κατευθυντηρίων γραμμών. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν μπορεί να τις καταλάβει ο μέσος δικαιούχος ή και μια αρμόδια αρχή η, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη και πολλές φορές όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που υποτίθεται ότι θα βοηθήσουν θεωρούνται ως νομοθεσία και ανοίγουν, ε, ε, οδηγούν σε περισσότερα ερωτηματικά. Μια άλλη εξίσου επικίνδυνη ιδέα που ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αλλά συζητείται όλο και περισσότερο ανοιχτά είναι να λυθεί το πρόβλημα αποδυναμώνοντας ή και καταργώντας το μοντέλο επιμερισμένης διαχείρισης. Πιστεύουν κάποιοι ότι αν ε, συγκεντροποιηθούμε και πάρουμε ε, το δικαίωμα συναπόφασης, ε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Από τις συζητήσεις συμπεραίνω ότι Αντί για μικροδιαχείριση και συγκεντροποίηση από την Κομισιόν, χρειάζεται πραγματική και γνήσια επικουρικότητα. Αυτή που δημιουργεί εμπιστοσύνη και επιτρέπει στην ε, Κομισιόν να ε, επιτρέψει με τη σειρά της τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι απλούστεροι κανόνες για τους δικαιούχους είναι λίγοι και κατά προτίμηση οι ίδιοι ε, που ισχύουν στο κράτος μέλος και την εθνική του νομοθεσία. Ως ομάδα υψηλού επίπεδου προσπαθήσαμε να δείξουμε πώς ένα τέτοιο απλό μοντέλο ε, μπορεί να είναι. Καταρχήν να μιλήσω για τις προτάσεις της ομάδας και τι έκανε η Κομισιόν μέχρι τώρα στα πλαίσια της περίοδου 2014-2020. Η υλοποίηση έχει ήδη αρχίσει. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί με αλλαγές για να μην υπονομεύσουν τη σταθερότητα των κανόνων αυτές. Όμως είμαστε ριζοσπάστες σε τομείς όπου η αλλαγή ήταν δυνατή και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. μας, οι ιδέες μας τώρα για μετά το 2020 και θα γιατί θα δείτε γραπτός συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια των συστάσεών μας όταν οριστικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί ε, θα ε, δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι προτείνουμε. Τώρα, για την περίοδο 2014-2020 θα γνωρίζετε ότι ε, εγκρίναμε έξι εκθέσεις για διάφορες περιφέρειες, ε, απλές λύσεις που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απλουστευμένα κόστη, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υπερθεματισμός, έλεγχος θα πω ορισμένα πράγματα. Η σταθερότητα των κανόνων είναι πολύ σημαντική. Ε, παίρνει χρόνο για να έχουμε συστήματα και ε, εργαλεία ε, τεχνολογίας της πληροφορίας. Αν ε, αλλάζουν οι κανόνες κάθε 7 χρόνια και με τις καθυστερήσεις που συμβαίνουν πάντα τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν μπορούν απόλυτα να αξιοποιηθούν, και έτσι θα, δεν θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα πλούστευσης... ε, τότε χάνουμε πολύ. Επίσης, ε, ο κανονιστικός υπερθεματισμός ε, ε, είναι ένας κίνδυνος. Είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Ε, πρέπει όμως να υπάρξει εμπιστοσύνη στα κρατη που θα δίνουν τα κονδύλια. Πολλές φορές οι στάσεις μας δεν είναι νομοθετικές. Πολλές φορές η αλλαγή των κανόνων σε αυτό το στάδιο της υλοποίησης ε, δημιουργεί ένα ρίσκο σύγχυση και καθυστερήσεων. Πιστεύουμε όμως ότι κάποιες νομοθετικές αλλαγές παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν. Είμαι ευγνώμων στην ε, Κομισιόν, διότι το Omnibus, το πολυνομοσχέδιο αυτό, συμπεριλαμβάνει πολλές προτάσεις που συστήσαμε. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πλουστευμένων δαπανών η πρόταση είναι πολύ καλή. Να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή Ρέτζι που υποστήριξε τις σημαντικές αυτές προτάσεις. Ελπίζω ότι η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, το Omnibus, θα οριστικοποιηθεί σύντομα, ούτως ώστε οι δικαιούχοι να αρχίσουν να, να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και εκτίμησα μια ε, πρόσφατη έκθεση της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής Ρέτζη σχετικά με τα δομικά στοιχεία της Επιτροπής Συνοχής. Μιας πολιτικής που περιλαμβάνει πολλές ιδέες και μιας έκθεσης που περιλαμβάνει πολλές παρόμοιες ιδέες με τις δικές μας. Για τον έλεγχο είχαμε πολλές προτάσεις ε, μη νομοθετικές που πρέπει όμως να ε, εφαρμοστούν. Πολλοί είχαν εμπειρία από τον έλεγχο στην περίοδο 2014-2020. Οι περισσότερε καταγγελίες προέρχονται από τους προηγούμενους κανόνες. Αλλά εγώ είμαι ευγνώμων στου ελεγκτές της Επιτροπής που έδωσαν σοβαρή συνέχεια το αίτημά μας για μεγαλύτερη ε, εμπλοκή στο σύστημα της ε, υλοποίησης. Κάποιοι ελεγκτές θεωρούν ότι αυτό θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι αυτό χρειάζεται για να προλάβουμε τις ε, διορθώσεις και να μειώσουμε τις διαφωνίες. Προσβλέπω στα αποτελέσματα του έργου των ελεγκτών που θα βοηθήσουν στη μείωση του κανονικού υπερθεματισμού. Ε, τώρα αξιοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές τους ελέγχους από άλλα προγράμματα και έτσι θα ε, ε, απαλληφθούν άσκοπες διαδικασίες. Μετά το 2020 πιστεύουμε ότι περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν. Την τελευταία δεκαετία τα ταμεία αυτά επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη των περιφερειών. Αυτό εν μέρη επετεύχθη ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των ε, επενδύσεων της Ένωσης ε, για την, ε, τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις καλύτερες κρατικές δημόσιες συμβάσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια, όλο και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι έχουν προστεθεί. αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου τα θετικά αποτελέσματα επισκιάζονται και τα ταμεία ε, επικρίνονται δυσανάλογα για σφάλματα στις δαπάνες και για ορισμένα παραδείγματα ε, απατών. Μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο να αντιμετωπίσουμε τις επικρίσεις και να απαλείψουμε τα σφάλματα, τα οποία ήταν μικρά, ενώ αντιμετωπίστηκαν με πάρα πολλούς κανόνες, που αντί να βοηθήσουν, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα των περιφερειακών ε, διοικήσεων και των δικαιούχων να διαχειριστούν με σόφρονα και αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια. Ε, πολύ λιγότεροι κανόνε. Αυτή είναι μια πρώτη προτεραιότητα για την περίοδο μετά το 2020. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα πάντα. Για πολλέ διατάξει είναι καλύτερα να επιμείνουμε, να αφήσουμε την τωρινή διατύπωση, διότι οποιαδήποτε νέα διατύπωση θα, θα υπονόμευε την κοινή ε, ερμηνεία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύουμε ότι αντί να επανασχεδιάζουμε το σύστημα κάθε ετία... όπως γίνεται τώρα, για το θεσμικό πλαίσιο περνάμε σε μία μόνιμη προσέγγιση που δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο όπως γίνεται τώρα για τους κανόνες ε, που υπάρχουν στον δημοσιονομικό κανονισμό. Πρώτα όμως θα πρέπει να πλουστεύσουμε ριζικά ή να απαλείψουμε αυτά που έχουμε. Για παράδειγμα, για έργα που δημιουργούν έσοδα, τη γεωγραφική ε, επιλεξιμότητα, τα ε, δημοσιονομικά ε, ε, μέσα. Αυτά είναι τα πρώτα. Δεν θα πρέπει να επιστρέψουν μεταμφιεσμένα ως κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμοί. Μόνο αυτοί οι κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν στον κανονισμό επιτρέπονται, ούτως ώστε να μπορεί ο νομοθέτης να παρακολουθεί και να έχει υποέλεγχο αυτή τη διαδικασία. Δεύτερο μεγάλο θέμα, πλήρης ευθυγράμμιση των οριζοντίων κανόνων, όπως κρατικές ενισχύσεις. Ε, ε, ένα πρόβλημα προέρχεται από κανονισμούς που δεν υπάρχουν στο κανονισμό για τη συνοχή. Το Horizon 2020 ή το EFSI, το Ταμείο για τις ε, Στρατηγικές Επενδύσεις, έχουν βρει διαθέσιμες λύσεις για τους δικαιούχους. Εμείς το 2000, για την περίοδο 2014-2020 ζητήσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και το επαναλαμβάνουμε ε, έντονα και για το μέλλον. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης, με τον ίδιο τρόπο τα έργα. Τέλος, έλεγχη ε, και λογιστική έλεγχη, εσωτερική έλεγχη. Αν δούμε τις στατιστικές, βλέπουμε ότι τα περισσότερα έργα ποτέ δεν θα υπόκεινται σε έλεγχο που θα καλύπτεται με τις, από τις αρχές αυτές. Κατά μέσον όρο, λιγότερο από 3% των ε, ε, πράξεων ελέγχονται από τους ελεγκτές. Είναι σαφές ότι όταν υπάρχουν παράπονα για τους ελέγχους, τις συγχαίουν με τις επαληθεύσεις της διαχείρισης που ισχύουν για το 100% των έργων ή άλλων ελέγχων από τις ε, αρμόδιες αρχές. Η έλεγχη ε, αυτή είναι λιγότερο επαχθής, με λιγότερους κανόνες θα ε, προχωρήσουν πολύ στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σε άλλους τομείς. Όταν ζητάμε από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές να ε, κάνουν πάλι ό,τι έχει γίνει από άλλους αρμόδιους φορείς, τότε η επικάλυψη είναι αναπόφευκτη. Και περνώ στο τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω σήμερα, η διαφοροποιημένη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να βασίζεται στην ποσότητα των κονδυλίων ε, για ένα έργο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η πραγματική αναγνώριση της επικουρικότητας. Ε, θα πρέπει να είναι κάθε έργο ανοιχτό σε όλους, ακόμα κι αν στην αρχή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεν θα πρέπει να ε, ορίζουμε κάθε επιλογή σε ενωσιακό επίπεδο. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι για τα κονδύλια και όχι μόνο στα πλαίσια του ενωσιακού προϋπολογισμού. Θέλουμε ένα σύστημα όπου τα κονδύλια θα δίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και θα ελέγχονται από τους εθνικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα. Η βασική αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και της Κομισιόν σε ένα τέτοιο σύστημα θα επικέντρωνε στα παραδοτέα συγκεκριμένες βελτιώσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ε, όπου θα γίνονται πληρωμές. Μια τέτοια ε, απλούστευση βάσει της επικουρικότητας δεν θα μείωνε τη λογοδοσία αλλά θα έδινε τη δυνατότητα αποτελεσματικότερων ελέγχων σε περισσότερα κράτη-μέλη και περιφέρειες και θα αύξανε την εμπιστοσύνη προς την Κομισιόν και στα κράτη-μέλη απελευθερώνοντας πόρους που τώρα δαπανώνται για ελέγχους άσκοπων ε, καθηκόντων. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, για αξιόπιστη δαπάνη αυτό θα οδηγούσε σε άμεσα ωφέλη και τώρα και στην επόμενη περίοδο. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα της τωρινή νομοθεσίας για να είναι λιγότερο περίπλοκη. Ε, αυτό θα ε, δημιουργούσε ένα σταθερό πλαίσιο και θα μπορούσαν και άλλοι να ε, επιταχύνουν για να πληρούν και εκείνοι στο μέλλον τις προϋποθέσεις θα, τελειώσω, θα ολοκληρώσω με τα συμπεράσματα για μετά το 2020 τις επόμενες εβδομάδες. Ε, για τα ΕΔΕΤ ένα σύστημα μπορεί να είναι απλό και αποτελεσματικό. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Ε, ελπίζω κυρία Πρόεδρε ότι θα παρευρεθείτε στις 11 Ιουλίου στην τελευταία μας συνεδρίαση όπου θα συζητήσουμε τις συστάσεις. Στα πλαίσια του μετά του 2020 οι ε, νομοθέτες θα πρέπει να ε, φροντίσουν ώστε η πρόταση για την απλούστευση να μην υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήδη στην αρχή της εργασίας της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου, δικός μας εκπρόσωπος ήρθε για να σας ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο σας. Οπότε, μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, συνάδελφοι, ερωτήσεις. Η κυρία Κρέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Κάλλας για την έκθεση αυτή. Εγώ είμαι υπεύθυνη εισηγήτρια για το πολυνομοσχέδιο, για τη διαδικασία Omnibus στην Επιτροπή αυτή και όπως είπατε για την περίοδο 2014-2020 ε, στη διαδικασία Omnibus για την πολιτική συνοχής έχουμε πολλές καλές προτάσεις. Τις έχουμε συμφωνήσει ήδη. Στην έκθεση μου βέβαια εστίασα στην αλλαγή για την πολιτική συνοχή. Και στο δημοσιονομικό κανονισμό ό,τι άμεσα έχει σχέση με αυτό. Στο Στρασβούργο είχαμε μια συνάντηση ε, που την, κάλεσε, τη συγκάλεσε η κυρία Γκρέσλε που είναι η κύρια εισηγήτρια και εξεπλάγει λίγο διότι η κυρία Γκρέσλε ξεκαθάρισε εκεί ότι δεν μπορεί να πει αν η αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού θα επιφέρει ωφέλη ή όχι. Φοβάται δηλαδή ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγχυση και οι υπάλληλοι της Κομισιόν δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν βράχει πρόθεσμα τη, τη, τον καινούριο κανονισμό. Ούτε θα ανταποκριθούν ε, όσοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των έργων με βάση το δημοσιονομικό κανονισμό των τωρινών Μου έκανε εντύπωση γιατί νόμιζα ότι η απλούστευση ε, είχε μεγάλο νόημα και ήταν πολύ θετική. Εσύ πώς το Εσείς πώς το εκτιμάτε αυτό. Γενικά για τον προϋπολογισμό. Διότι πρόκειται για μία άρδιν αλλαγή νομοθετική. Μια αλλαγή σε βάθος. Έχετε ε, κάποια άποψη για το αν αυτό θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα ή αν ενδεχομένως θα δημιουργήσει μεγαλύτερο χάος από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάλετιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας που μας παρουσιάσατε το έργο σας μέχρι τώρα και τι προτείνετε για το μέλλον. Χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη και αυτό ξανά και ξανά στην παρουσίασή σας. Γιατί όντω πρόκειται για θέμα εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Επιτροπή και τι χώρε μέλη και μετά βέβαια και μέσα στι χώρε μέλη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί πράγματι. Και τώρα που αναφερθήκατε στις 5.000 σελίδες κατευθυντήριες γραμμές, ε, δεν ξέρω ότι κατά πόσο πολλές ε, διαχειριστικές αρχές αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων αυτών ε, γραμμών και τι περιλαμβάνουν όσον αφορά την διαχείριση. Τώρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα αναπτύξουμε περισσότερο την ηλεκτρονική συνοχή όχι μόνο μεταξύ χωρών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μέσα στην κάθε χώρα μέλος. Έτσι ώστε ο τελικός δικαιούχος να μην πρέπει να στέλνει κάθε χαρτί, αντίγραφο κλπ. στην εφαρμοστική αρχή αλλά να υπάρχει τρόπος να παρακολουθούμε τα προγράμματα μέσα στο σύστημα. Και αυτό που είπατε για την απλοποίηση. Τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος με το Omnibus, προτείνονται αλλαγές στον κανονισμό, αλλά και πάλι έχουμε ελεγκτές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν inputs και όχι outputs για το απλοποιημένο κόστος και συνήθως επικεντρωνόμαστε στο input και γι' αυτό και δεν μπορούμε να αλλάξουμε και να εφαρμόσουμε απλοποιημένες εναλλακτικές κόστους. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε και την οτρυπία. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φαν Μίλντεμπορκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Κάλλας για την παρουσίασή σας. Συγχαρητήρια και σε εσά και στα άλλα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου. Έχω μερικές ερωτήσεις, γιατί πολύ χάρηκα που άκουσα ότι και εσείς θέλετε περισσότερη σταθερότητα. Συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω και εγώ ότι δεν είναι σοφό κάθε θητεία να αλλάζουν όλοι οι κανόνες. Όχι. Χρειαζόμαστε κάποιο βαθμό προβλεψιμότητας, σταθερότητας και τη προγραμματική περίοδο και στην απορρόφηση των κονδυλίων. Όταν ερχόμαστε τώρα στις επαληθεύσεις, έλεγχο και διαχείριση, συμφωνώ με το ενιαίο σύστημα, αλλά από ό,τι φαίνεται συζητήσατε και για κάποια διαφοροποίηση. Συζητήσατε τα κριτήρια, το πεδίο εφαρμογή μπορείτε να μας πείτε περισσότερα επί του θέματος. Θα ήταν εφικτό στο μέλλον να έχουμε διαφορετικούς ελέγχους και ελεκτικά συστήματα στις διάφορες χώρες ανάλογα με τις επιδόσεις τους, όσον αφορά δηλαδή την ορθή απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση μου. Δεύτερον, συζητάμε πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συνέργειες. Εσείς θα συμπεριλάβατε στις τελικές σας συστάσεις πώς να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα διευθυντικά ταμεία αφενός και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon 2020 και άλλα γιατί πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο. Και τέλος, ποια θα ήταν η σύστασή σας για πιο αποτελεσματική επιμερισμένη διαχείριση, στην πράξη δηλαδή, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, ποιες είναι οι συστάσεις σας. Ρωτάω δηλαδή, θα έπρεπε να ενισχύσουμε περισσότερο την αρχή της εταιρικής σχέσης Χρειαζόμαστε έναν πιο λεπτομερή κώδικα διοντολογίας, μήπως. Τι θα είχατε να συστήσετε. Ευχαριστούμε κυρία Διαμάτου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο κύριο Κάλλας για την παρουσία του. Ασχολείται με τα θέματα αυτά της απλοποίησης από τον Οκτώβριο του 2015 εμείς γνωρίζουμε τις συστάσεις τις οποίες μας παρουσιάσατε και γι' αυτό θα θέσω δύο ερωτήσεις. Επί τη βάση της δικής σας εμπειρίας, τι πιστεύετε για την πρόταση δημιουργίας ε, εξάντε αιρεσιμότητας για την εταιρική σχέση και για την ε, εμπλοκή των διαφόρων ε, συμμετεχόντων εξ αρχής. Ξέρω ότι υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς που απαιτεί την υποχρεωτική συμμετοχή. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα οι εμπλεκόμενοι ότι η συμμετοχή τους μερικές φορές είναι μόνο τυπική. Εμείς προτείνουμε μία εκ των προτέρων λοιπόν ερεσιμότητα συγκεκριμένη με εκ των υστέρων έλεγχο. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει την συμμετοχή όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πολλές φορές νιώθουν περιφρονημένες από τις ίδιες τους τις κυβερνήσεις. Και δεύτερον, τι μπορείτε να μας πείτε περισσότερο για τους κανόνες λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Έχει γίνει αναφορά στην ενιοποίηση των κανόνων, διεύρυνση των επενδυτικών ε, Διαφορετικών ταμείων των πλεονεκτημάτων των προγραμμάτων που γίνεται ο αντικείμενο κεντρικής διαχείρισης. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Καλώς, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλλας να σας ευχαριστήσω εσάς που μας προσκαλέσατε και να ευχαριστήσω εκ νέου τον κύριο Κάλλας γιατί έχει οργανώσει μέχρι τώρα μια ιδιαίτερα ευφυή συζήτηση για το τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτό που μας ενδιαφέρει στο μέλλον. Έγιναν πολλές προτάσεις από πλευράς του κυρίου Κάλλας μετά από προτάσεις ε, της ε, ομάδας εργασίας που περιλαμβάνονται στην πρόταση Omnibus απλοποιημένο κόστος, μοναδικά ηλεκτρονική μορφή και πολλά είναι ακόμα τα θέματα στα οποία θα επανέλθουμε στο μέλλον. Για τους λογιστικούς ελέγχους υπάρχουν αρκετές προτάσεις από την ομάδα υψηλού επίπεδου που έγιναν δεκτές από τις ελεγκτικές τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές περιλαμβάνουν αυτό που είπε ο κ. Κάλλας για την εμπλοκή των ορκωτών λογιστών στην επικύρωση της λειτουργίας του προγράμματος ε, να πω ότι οι ελεγκτές θα πρέπει να βοηθούν τις αδειοδοτικές εξωτερικές υπηρεσίες να ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές και να τις πιστοποιούν. Θα απαιτήσει κάποιο χρόνο γιατί δεν είναι κάτι το οποίο κατέχουν, αλλά θα δουν όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος πώς θα απλοποιηθεί η διαδικασία. Και θα πρέπει να δούμε επίσης ε, και τι γίνεται με τις ε, αξιολογήσεις που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει οι ελεκτικές αρχές ε, να δουν τι κάνουν οι άλλες χώρες και να υιοθετούν τις χρήσιμες πρακτικές τους. Ήδη για το 2020 έχουμε δώσει εμείς λεπτομερείς απαντήσεις στην ομάδα υψηλού επίπεδου και για το μετά του 2020 όταν δείτε τις προτάσεις της Επιτροπής νομίζω ότι θα αντικατοπτρίζουν τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Συμμετέχουμε λοιπόν στην ομάδα υψηλού επίπεδου, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτά τα οποία μας προτείνουν, μερικές φορές μας βρίσκουν σύμφωνος, άλλες όχι, αλλά σίγουρα βοηθούν ιδιαίτερα την συζήτηση που γίνεται. Ευχαριστώ κύριε. Um, uh, okay. I think many interesting... Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Έχουμε στραφεί προς το μέλλον για το 2020, έχουμε επενδύσει αρκετά όμως και για το θέμα της πρότασης Omnibus. Έχουμε δημιουργήσει, θα έλεγα, επικοδομητικές προτάσεις για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον για το 2020 και μετά. Μία ερώτηση από πλευράς μου. Εγώ δεν περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει γρήγορα για τις προτάσεις για το μετά το 2020. Από ό,τι φαίνεται, ε, οι προτάσεις για μετά το 20 είναι ένα είδος ταμπού, το οποίο δεν συζητιέται. Εμείς όμως τα συζητάμε τα θέματα αυτά και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Κάλλας, το τι εσείς περιμένετε. Σας ευχαριστώ αγαπητά μέλη, ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Πραγματικά θίξατε πάρα πολλά και ευαίσθητα θέματα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, και αυτό αφορά και μένα, ότι εμείς ασχολούμαστε με την απλοποίηση των κανόνων υπέρ των ωφελουμένων και εμπλεκομένων σε σχέση με τις μορφές αυτές χρηματοδότησης από διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης των ταμείων αυτών. Και προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα οποία μαθαίνουμε λοιπόν στην έκθεσή μας. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τις λεπτομέρειες και τώρα μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με ευρύτερο τρόπο. δημοσιονομικός κανονισμός, σαν παράδειγμα. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Γκρέσλε, με την οποία συνεργαστήκαμε όταν ήμουν υπεύθυνος αντιπρόεδρος για τις απαλλαγές. Και αυτό το οποίο κάναμε ήταν να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ελέγχου των δαπανών. Επίσης θέσαμε άμεσα το θέμα του ποσοστού του επιτρεπόμενου λαθών για να το φέρουμε, να το χαμηλώσουμε σε ανακτά επίπεδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται ακόμα και τώρα ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο λαθών που δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου. Για το δημοσιονομικό κανονισμό λοιπόν η συζήτηση η οποία θα γίνει θα είναι πάρα πολύ θερμή. Η συζήτηση αυτή έγινε και για τα διαφθορτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στο παρελθόν ένας δημοσιονομικός κανονισμός είναι με μια βασική ιδέα, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ ε, και από εσά. έτσι ώστε να δούμε πράγματι ε, πού πρόκειται να καταλήξει η διαδικασία αυτή. Να υπογραμμίσω επίσης ότι από τη μία υπάρχει μια σειρά χωρών οι οποίες χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι καθαροί συνεισφορείς και θέλουν φυσικά οι δαπάνες να γίνονται αντικείμενο τέλειας διαχείρισης. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Θέλουν να υπάρχει, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη χαλαρότητα και υπάρχουν και ε, ανώτατοι υπαλλήλοι στις διαχειριστικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι ε, φοβούνται ότι θα κάνουν λάθη βέβαια και γι' αυτό υπογράμμισα το θέμα της εμπιστοσύνης. Πάντως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και ανοχή για τους κινδύνους αυτούς δεν έχουμε καταλήξει ακόμα βέβαια σε ένα ξεκάθαρο ποσοστό αποδοχής ε, για τα λάθη, γιατί είναι πολύ πολιτικό το θέμα, όπως και άλλα θέματα τα οποία θέσατε, όπως η κοινή διαχείριση. Πώς θα λειτουργήσει η κοινή διαχείριση δεν είναι θέμα μαθηματική, είναι θέμα ισορροπίας ανάμεσα στις συγκεντρωτικές λήψεις αποφάσεων και τις μεμονωμένες εθνικές και σχετικά επίσης και με τα θέματα των διαφοροποιήσεων θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ένα συναδελφό σας ότι και στη δική μας ομάδα το θέμα το συζητάμε Προσπαθούμε να συλλέγουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής μέχρι τώρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με μεγαλύτερο πνεύμα εμπιστοσύνης από ό,τι μέχρι τώρα. In Προσπαθούμε όμως αυτή την διαφοροποίηση. Ε, σαν παράδειγμα υπάρχουν κάποια μέλη και στην Αυστρία τα οποία έχουν κάνει προτάσεις για το πώς θα γίνει και εδώ εμείς προτείνουμε σαν ομάδα υψηλού επίπεδου Η πρόταση αυτή δεν θα πρέπει να μην συνοδεύεται από κανόνες ε, οι οποίοι τελικά να βασίζονται και σε αριθμητικά ποσοστά γιατί ναι μεν ένα πράγμα είναι η αριθμή, αλλά βασικά το θέμα της εμπιστοσύνης είναι σημαντικό και γι' αυτό εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τον δημοσιονομικό σας κανονισμό. Ε, the to have uh, rules and, and... Εντάξει, όλοι θέλουμε ευκολότερους και απλούστερους κανόνες και διαφάνεια, αλλά τώρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που συζητήσαμε. Ακούσαμε πάρα πολλούς εμπλεκομένους, το συζητήσαμε και εμείς. Είναι κάτι το οποίο είναι σαφώς ε, που ξεχωρίζει είναι η ανάγκη για σταθερότητα. Αν δημιουργήσεις ένα σύστημα ε, και θέλεις ε, να το χρησιμοποιήσεις για να επενδύσεις σε ηλεκτρονικές λύσεις, δεν μπορείς να το αλλάζεις αυτό συνέχεια. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη, θέλει να πει ο μιλητής, επένδυση, και απαιτείται μια σταθερή λύση. Τίθεται θέμα σταθερότητας λοιπόν και υπάρχουν και διαφορετικά βέβαια σε διάφορες ε, χώρες επίπεδα κατάρτισης, ε, σε επίπεδο ελεγκτικών αρχών, αρχών εποπτείας και αυτοί που ωφελούνται οι δικαιούχοι δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι. ...παρόλα αυτά η δυνατότητα του e-government στην απλούστευση είναι στην απλοποίηση είναι τεράστιο και ήδη έχει γίνει σε ορισμένες χώρες μέλη μεταξύ των οποίων και την ειδική μου. και νομίζω ότι περιλαμβάνονται και στις προτάσεις της Επιτροπής. Το θέμα της σταθερότητας τώρα είναι κάτι το οποίο βοηθιέται ιδιαίτερα από το e-governance και η πρότασή μας να μειώσουμε τον αριθμό των θεμάτων ήταν κάτι το θετικό, αλλά μετά είδαμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με κατευθυντήριες γραμμές που φτάνουν 5 και 6 χιλιάδες σελίδες, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι' αυτό υπάρχει ουσιαστικά η ποσότητα αυτή είναι ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης ή ουδήποτε επίπεδου ελεγκτικών και εποπτικών αρχών. Και ανεξάρτητα λοιπόν τις επιπλέον καθευθυντήριες γραμμές, τις οποίες η επιπεδου ελεγκτικων και εποπτικων αρχων και ανεξαρτητα λοιπον Επιτροπή με χαρά μπορεί να παράγει συνεχώς, αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό, Our basic idea was και γι αυτό ακριβώς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις αυτές ε, κατάργησης ε, των κατευθυντήριων γραμμών. Από τη μία υπάρχουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις και πέραν τούτου δεν. Και το θέμα είναι βέβαια ποιος θα ερμηνεύσει ε, το αποτέλεσμα της εφαρμογής των ε, νόμων, των κανόνων, αλλά θα δούμε. Και όπως είπα, οι προτάσεις που κάνουμε μειώνουν ριζικά τον αριθμό των κατευθυντήριων προτάσεων της Επιτροπής και των αρχών ελέγχου και κάποιες υποτίθεται πλευρές, κάποιοι τομείς δεν είναι εύκολο να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης χωρίς. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε εν πολλής κάποιες κατευθυντήριες να μην τις έχουμε μπροστά μας. Ενδιαφέρον επίσης και το θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Μίλτεμπεργκ για τα διαφορετικά ταμεία και τους διαφορετικούς κανόνες. Όταν είναι ένας μια μικρή μεσαία επιχείρηση είναι δικαιούχος και να, ζητά να χρηματοδοτηθεί από διάφορες πλευρές, από περιφερειακά ταμεία και από το Horizon 2020 και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μορφών χρηματοδότησης. Εμείς λοιπόν αυτό που προτείνουμε σαν ομάδα προς την Επιτροπή είναι στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας να δει πώς μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Ε, και φυσικά τίθεται το θέμα αυτό, το οποίο όμως και με πολιτικούς όρους, τίθεται και με πολιτικούς όρους. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Πάντως σε επίπεδο διαδικασιών νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση. Λοιπόν, το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν μία χώρα με ένα σετ κανόνων μόνο. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και δεν θα το πετύχουμε εύκολα. Τώρα για την εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι είναι σαφής η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι εξ ονόματος της Επιτροπής. Εγώ ήμουν υπεύθυνο για την απαλλαγή στον προϋπολογισμό και νομίζω ότι θα σαφώς και πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ είχα προτείνει οι αποφάσεις ε, να λαμβάνονται με ξεκάθαρο τρόπο έτσι ώστε να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά ένας συνάδελφος που είναι υπεύθυνος για θέματα υγείας είπε και τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Τώρα ξαφνικά απέκτησα 60 εταίρους. Τι θα κάνουμε όλους αυτούς. Πώς θα πάρω αποφάσεις όταν έχω 60 παριστάμενους που θέλουν να πάρουν μέρος στην απόφαση. Και ποιος είναι ο πιο σημαντικός, ποιος είναι ο λιγότερο σημαντικός ε, που πολλές φορές μεταξύ τους τσακώνονται και όλας και δεν ξέρω τι να κάνω. Σύνεπως λοιπόν είναι ε, μια ευθύνη που άπτεται της λήψης απόφασης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς ισόρροπα δηλαδή το θέμα δεν μπορεί να είναι αυστηρά ποσοτικός, αριθμητικός. Εάν τώρα ένας που λαμβάνει αποφάσεις μπορεί σοβαρά να κατηγορηθεί ότι αγνοεί την κοινωνία των πολιτών και τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών, αυτό είναι φυσικά κάτι το πάρα πολύ κακό. Από την άλλη όμως, θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να προσπαθήσει να ασκήσει την επιρροή της με ισόρροπο τρόπο και υπάρχουν πολλά μέλη στην ομάδα μας τα οποία σαν παράδειγμα για τις ε, παρεμβάσεις στον τομέα των ε, πόλεων, της πολιτικής για τις ε, πόλεις ζητούν να υπάρξει μια ισορροπημένη συνεργασία. Και τώρα η σχέση ανάμεσα στην συγκεντρωτική διαχείριση και την αποκοινού διαχείριση. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις <clears throat> να καταργηθεί η αποκοινού διαχείριση και να υπάρχουν μόνο συγκεντρωτικές λήψεις αποφάσεων. Και πράγματι σε κάποιους τομείς όπως οι μεγάλες υποδομές, κοινέ υποδομές, αυτό έχει και λογική πολύ μεγάλα προγράμματα, πολύ μεγάλα έργα, πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλές χώρες, οπότε είναι καλύτερο να υπάρχει μια συγκεντρωτική μορφή διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο. Αλλά από την άλλη όμως και έρχομαι εδώ στην αποκοινού διαχείριση είναι μια μορφή γνήσιας επικουρικότητας και υπάρχουν μέλη της ομάδας μας που υπογραμμίζουν ότι απαιτείται να αναπτυχθεί η γνήσια αυτή από κοινού διαχείριση και ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές διαχειριστικές αρχές. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτές λοιπόν είναι όλες παρατηρήσεις τις οποίες κάνω και σκέψεις Καταλαβαίνετε ότι η ομάδα μας είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μεν, αλλά δεν ξέρω, ίσως και οι ιδέες μας να μην επαρκούν. Πάνω προσπαθούμε να εκθέσουμε τις απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος και εγώ σαν τέος πολιτικός μπορώ να πω είναι ότι οι προτάσεις που έχουμε κάνει είναι χρήσιμες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο και για όλους όσους συμμετέχουν. Ευχαριστούμε κύριε Κάλλας εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δώσατε, για την αρχική σας παρουσίαση βέβαια και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην τελευταία σας αυτή συνάντηση. Ευχαριστούμε για το έργο σας επίσης. Συνεπώς μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε. Βασικά κλείνει το ανοιχτό τμήμα της συνεδρίασής μας και ζητάω από τους συντονιστές, παρακαλώ, να παραμείνουν για να συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών. Συμφωνούν οι συντονιστές?